Okay. I think we can start. Να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση με μια δημόσια ακρόαση με την Έλκη Κένι. Καλώς την κυρία Κένι. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας, στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου, αλλά είναι η πρώτη στη δική μου προεδρία. Προεδρία ως γυναίκας Προεδρού. Καλώς ήρθατε και πάλι να πω ότι πραγματικά χαιρόμαστε για την καλή μας συνεργασία που έρχεστε όποτε χρειάζεται για αυτές τις επίσημες ακροάσεις και για άλλες ε, συνεννοήσεις που είχαμε ως τώρα. Η δημόσια ακροάση βασίζεται στο πλαίσιο του κανονισμού για τον νέο μηχανισμό ε, εξηγένσης και το νέο ε, συμβούλιο ε, και τις πρακτικές που επικρατούν για τη δημοκρατική λιγοδοσία και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο νέο, στο νέο Συμβούλιο εξηγένση. Βάσει των ε, τακτικής διαδικασίας θα έχουμε την ενεκτή ομιλία τη κυρία Κέρνη για 10 λεπτά με ε, ένα ερωταπαντήσεων 5 λεπτών. Κυρία και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που μπορώ ε, δημοσίως να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Νομίζω ότι έχουμε κοινά συμφέροντα να φροντίσουμε να είναι όσο γίνεται πιο ισχυρός και αποτελεσματικός ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης και στην εισήγησή μου θα ε, σας περιγράψω τους τομείς προτεραιότητας και κατόπιν θα σας περιγράψω τις προτεραιότητες μας για το 2020, διότι έρχεται σύντομα το 2020. Λίγα λόγια για τη δέσμη μέτρων για, την, για τις τράπεζες. Η εφαρμογή αυτής της δέσμης μέτρων θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα για μας τους επόμενους μήνες και αυτό δεν αληθεύει απόλυτη. Ήταν ήδη σημαντική προτεραιότητα για μας και τους τελευταίους μήνες. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε και περνάω στο BRRD1, ε, τον ε, κύκλο σχεδιασμού 2018-2019, ε, όπου είχαμε εφαρμόσει μία προσέγγιση σε στάδια. Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς θα έχουν σχεδόν όλες οι τράπεζες δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Έχουμε όμως κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή και θα ε, ε, σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Οι δέσμοι μέτρων αναφέρεται σε απαιτήσει για την απορρόφηση ε, ζημιών που έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και είναι αυτή η απέτηση και τώρα περιπλέκονται τα πράγματα, ισχύει ήδη για συστημικές τράπεζες παγκοσμίω και ευθυγραμμίζει το πλαίσιο ε, ε, ε, για τις ελάχιστες απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Οι συστημικές τράπεζες και οι τράπεζες με στοιχεία του ενεργητικού που ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια, καθώς και οι θα πρέπει να έχουν σε δευτερεύοντα ομόλογα, δευτερογενή ομόλογα, ε, τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Οι άλλες τράπεζες θα πρέπει ούτω ή άλλω να αξιολογηθούν και ε, το ε, ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να απαιτήσει κάτι παρόμοιο για τις τράπεζες αυτές. Ας έχουμε κατά νου ότι όλες οι τράπεζες και όχι μόνο οι πολύ ε, μεγάλες ε, θα πρέπει να ε, εξηγιανθούν και οι ελάχιστες απαιτήσει είναι τμήμα της προσπάθειας αυτές. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε από ατομικές απαιτήσει σε εσωτερικές απαιτήσει. Αυτό μπορεί να το θεωρήσετε ε, τεχνικό ζήτημα, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό οι θηγατρικές ε, θα πρέπει να εκδίδουν ε, χρηματοπιστωτικά μέσα και να είναι υπόλογες στις στις μητρικές οντότητες. Θα σταματήσω τότε ότι παραγίνονται τεχνικά τα πράγματα, αλλά πάντω οι ελάχιστε απαιτήσει είναι ε, μάλλον η σημαντικότερη προϋπόθεση για την εξυγίανση των τραπεζών, η εξασφάλιση δηλαδή ε, επαρκών ε, κεφαλαίων ε, για να απορροφηθούν οι ζημιές και έτσι ε, αντικαθίσταται η διάσωση με πόρου των φορολογουμένων από ιδιωτικό φορέα. Ε, έχουμε πολυετή προσέγγιση στις ελάχιστες απαιτήσει με στόχο να διατηρήσουμε την αναλογικότητα του συστήματος, ε, διατηρώντας ταυτόχρονα και συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και διατηρώντας ε, υψηλά πρότυπα σε όλη την Τραπεζική Ένωση. Και σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό και τα επόμενα χρόνια. Η έλλειψη επαρκών MRL μπορεί να μας ε, εμποδίσει από το να έχουμε την προτιμητέα ε, στρατηγική εξυγίανση. Ε, θα σας δώσουμε στοιχεία συνολικά, αλλά να γνωρίζετε ότι τα μεγέθη αυτά περιγράφουν όσους έχουν επαρκή Μαριέλη και όσους έχουν λήψεις. Πάντως 25,2% της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο αντιπροσωπεύουν τα Μαριέλη, ενώ συνολικά για το σύνολο των τραπεζών που αξιολογήσαμε ανέρχεται σε 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2018 που αντιστοιχεί σε ανάλογα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Για τις τράπεζες όπου δεν υπάρχουν υποχρεωτικές απαιτήσει. Αναμένουμε κατά μέσο όρο 17,8% των ε, στοιχείων του ενεργητικού που θα πρέπει να αντικατασταθούν από δευτερογενή ε, μέσα. Ε, η μέση έλλειψη MREL, μέσος όρος, είναι το 2% των στοιχείων του ενεργητικού, των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού. Ε, περίπου 140 ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του προηγούμενου έτους. Τώρα με τις νέες απαιτήσει θα αλλάξουν τα νούμερα. Θα δούμε λοιπόν περισσότερες απαιτήσει, κάποια ενίσχυση, αλλά είναι ακόμα σημαντικό ο αριθμός όταν το συγκρίνουμε με τους δικούς μας πόρους. Και Πρέπει να σκεφτούμε ότι πέρσι ε, το 140 ε, εκδόθηκαν Εμαριέλ ε, ύψους 140 εκατομμυρίων και αυτό δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταφέρει ο τραπεζικός τομέας σε βάθος χρόνου. Και ζητώ συγγνώμη για το κρυολογήμά μου, λέει η ομιλήτρια. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στα θέματα από πλευράς πολιτικής. Ο ε, δεύτερος ε, ενίος μηχανισμός εξυγίανσης ε, θα τεθεί σε ισχύ τέλη του 2020 και έχουμε εργαστεί σκληρά για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας ώστε να είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή. Θέλουμε να είναι έτοιμη η νέα πολιτική Εμαριέλ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και να έχει γίνει και διαβούλευση με τον τραπεζικό τομέα σε κάποιους τομείς. Έτσι θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής του 2020 να αρχίσουμε συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ε, αυτό και να ε, να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ε, το πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπου θα ισχύει πια το SRM2 εφόσον ε, και τα κράτη-μέλη θα έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Γίνονται, λοιπόν, ε, γίνεται πολλή δουλειά, αλλά μπορεί να μην είναι ε, όλα πολύ εύκολα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές αλλαγές και επικεντρώνομαι τώρα στις ελάχιστες απαιτήσει. Χρειαζόμαστε πιο σαφείς προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα, δεύτερον μεγαλύτερη εξασφάλιση και τις εσωτερικές ελάχιστες απαιτήσει, ιδιαίτερα εντός των ομίλων, ε, για να γνωρίζουμε ποιοι μπορεί να κατέχουν ε, τα εσωτερικά MRL. Ε, πρέπει να πούμε όμως ότι η νέα νομοθεσία είναι ιδιαίτερος πολύπλοκη. Άλλωστε αποτελεί αντικείμενο ενός καλού συμβιβασμού. Ε, βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, το EBA, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις προκλήσεις. Οι πρόσφατες εμπειρίες μας μας δείχνουν ότι θα είναι αναπόφευκτο ε, το ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επιληθούν ε, θέματα εφαρμογής και αυτό είναι άλλο ένα επιχείρημα για την βαθμιαία εισαγωγή του νέου πλαισίου, διότι ήδη τώρα είναι σαφές ότι θα καθυστερήσει το δεύτερο επίπεδο. Θα πρέπει να ληφθούν δηλαδή οι πρώτοι θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρώτο στάδιο προτού να έχουμε την ε, τελική ε, απάντηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ε, και μια τελευταία παρατήρηση πριν προχωρήσω σε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μες. Είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης. Εδώ γίνονται παράλληλα διάφορες εργασίες. Πρώτον μπορεί να έχετε δει ότι έχουμε δημοσιεύσει τις προσδοκίες μας από τις τράπεζες, ένα έγγραφο δημόσια διαβούλευση μέχρι Αυτό το έγγραφο δεν περιέχει μια νέα σειρά πολιτικών. Ε, περιγράφει σε ένα ενιαίο έγγραφο τι περιμένουμε να κάνουν οι τράπεζες ώστε να ε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξυγίανσης. Ε, προσανατολισμός, κατευθυντήριες γραμμές, benchmarking, ώστε να έχει ο τραπεζικός τομέας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και για τις δικές μας αξιολογήσεις. Το έγγραφο αυτό, λοιπόν, ε, συμπληρώνει τα, τις λεγόμενες ε, επιστολές προτεραιοτήτων ε, που περιγράφουν τις προτεραιότητες για κάθε τράπεζα εντός ενός συγκεκριμένου έτους. Έτσι λοιπόν είναι προσαρμοσμένες οι προτεραιότητες αυτές σε κάθε τράπεζα και τους ζητάμε να ασχοληθούν με αυτέ ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο εξυγίανση. Παρέχουμε σαφή προσανατολισμό με συγκεκριμένα καθήκοντα και κατόπιν ε, ακολουθεί η αξιολόγηση του ενιαίου συμβολίου εξυγίανση, λίγο σαν σχολικό έλεγχο ε, όπου τους λέμε ε, πού θα πρέπει να επικεντρωθούν για να βελτιωθούν. Και με αυτή τη βάση, αν χρειαστεί, θα ξεκινήσουμε διαδικασίες ε, για τις τράπεζες που δεν έχουν λάβει το μήνυμα και δεν σημειώνουν παρκή πρόοδο. Πάντως, ε, νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο και πολύ ευχαρίστω θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, προβλέπουμε κάτι ακόμη έχουμε έναν χάρτη ε, όπου ε, καταχωρίζονται οι τράπεζες ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκονται στον στόχο της εξυγίανσης. Είχαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ε, όπου αναφερθήκαμε στις ε, αποχρώσεις του κίτρινου και του κόκκινου, του πορτοκαλί και του κόκκινου ε, αν σκεφτούμε ένα σύστημα σαν φανάρι του δρόμου. Όλα αυτά στόχο έχουν να βελτιώσουν τις δυνατότητες εξυγίανσης. Ένα θέμα πριν κλείσω ε, έχουμε μάθει πολλά και από προηγούμενες ε, αποφάσεις μας να μην ε, γίνει η εξυγίανση κάποιων τραπεζών. Θα θυμάστε ότι τον Αύγουστο αποφασίσαμε για μια πολύ μικρή τράπεζα που χρεοκοπούσε ήταν έτοιμη να ε, ε, χρεοκοπήσει ότι δεν ήταν προς ε, γενικό συμφέρον να διασώσουμε την τράπεζα αυτή και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να διαπιστώσουμε την περιγραφή αυτή για την αφαιρέγγια τράπεζα στην πράξη. Ένα τομεί όπου απαιτείται βελτίωση είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση ε, εξυγίανση και αφαιρεγγιότητα ε, συμπεριλαμβανομένου ενός καθεστώτος για την ε, ρευτοποίηση μιας τράπεζας που να συμπεριλαμβάνει και εναρμονισμένες διαδικασίες για την ανάκληση της άδεια. Αυτό εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση ε, την Εθνική Νομοθεσία. Πολύ ευχαρίστω, θα σας εξηγήσω περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό. Τέλος, τι έχουμε ακόμη στο θεματολόγιο μας. Ε, κάποια από αυτά είναι αρκετά γνωστά θέματα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία πάνω στον ε, τρίτο και, τελικό τελευταίο πυλώνα της τραπεζικής έντοσης. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια πολύ θετική ορμή γύρω από ένα ευρωπαϊκό καθεστώς διασφάλισης των καταθέσεων ε, και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί εντός της ε, παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Ε, δεν περιμένω να γίνει αυτό μέσα σε ένα έτος. Επίσης, θέλουμε ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Η πιο ισχυρή κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη είναι προς συμφέρον ε, όλων ε, και των, και επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και τέλος, ε, στον κατάλογο μου αυτόν, για να σας δώσω και τις τελευταίες ημερομηνίες, φυσικά, συγκεντρώνουμε πόρους για το Ταμείο Εξυγίανσης. Ελπίζουμε μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς να έχει ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Επίσης, όσον αφορά ε, την, ε, το backstop του ταμείου αυτού, ε, ελπίζουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύντομα. Ε, θα περιμένουμε άλλωστε και τα αποτελέσματα της αυριανής ε, συνεδρίασης του Eurogroup και θα έπρεπε να τα έχω πει τώρα αυτά με την ανάποδη σειρά. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε ακόμα κάποια λύση για την ρευστοποίηση. Ελπίζουμε το νέο έτος να φέρει νέες λύσεις. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και να επαναλάβω ότι δεσμευόμαστε να ασχοληθούμε με την εξυγίαση των τραπεζών. Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε πρώτα και την Τραπεζική Ένωση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ομιλήτρια, ξεκινώντας από τον κύριο Φέμπερ, το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Κιόνικ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, μετρική σας γλώσσα Ε, έχω βέβαια από, κάτι τελευταίο από μενέργεια που συνάχει, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Εδώ λοιπόν ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με το no credit was off, αυτή την αρχή, ότι κανένας πιστωτής δεν θα έχει χειρότερη μεταχείριση. Και τι γίνεται με, τις δική μας, ε, με το δικό μας σύστημα εθνικής εξυγίανσης σχετικά. για τις τράπεζες συνολικά έχουμε την ε, δυσκολία ότι δεν ξέρουμε πώς να ε, ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό και πότε. Και επίσης για αυτό το θέμα στο οποίο θα ενσκύψετε ξανά για το ευρωπαϊκό δίκαιο αφαιρεγγιότητας. Θα πρέπει και στο Συμβούλιο να συζητηθεί αυτό και ενδεχομένως να προχωρήσει και να γίνει παραδεκτό. Νομίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι που θα πρέπει να, να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Γιατί, όπως είπατε, εάν λάβουμε απόφαση αφαιρεγγιότητας, θα πρέπει να δούμε τι 19 διαφορετικέ απαντήσει που μπορεί να δοθούν για τι ε, περιπτώσει αφαιρεγγιότητας. Σε κάποιε χώρε υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα παράλληλα. Το άλλο επιχείρημα είναι αυτό που ανέφερα και εγώ, ότι δεν υπάρχει μία περίπτωση να πούμε ότι αν μια τράπεζα ε, υπάρχει περίπτωση να πτωχεύει και δεν είναι αρκετά μεγάλη για να περιληφθεί στο μηχανισμό εξυγίασης, μπορεί να μπει σε διαδικασία πτώχευσης και να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο από τη μια χώρα στην άλλη. Οπότε για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε. Η αφαιρεγγιότητα πρέπει να διασυνδεθεί με άλλες νομικές διαδικασίες και έχετε απόλυτο δίκιο. Εάν έπρεπε να ζητήσουμε ένα σύστημα αφαιρεγκαιότητα εναρμονισμένο. Δεν ξέρω αν θα παρακολουθούσαν τη συζήτηση όλοι ε, όσοι βρισκόνται σήμερα εδώ. Εγώ μάλλον θα έχω πάρει σύνταξη από καιρό. Το δικό μου επιχείρημα είναι όμως να είμαστε ταπεινόφρονε και να θεωρήσουμε ότι οι τράπεζες επτόχευση θα πρέπει να ρευστοποιηθούν και με ασφάλεια. Και τα επιχείρημα είναι να δούμε τι κάνουν και οι Αμερικανοί φίλοι μας, το FDIC. Ε, όπου διοικητικά τη ρευστοποίηση την αναλαμβάνει κεντρικά η τράπεζα με ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Και υπάρχει ε, μια αποτελεσματική διοικητική διαδικασία ταυτόχρονα. Αυτό θα ήταν μια ενδεχόμενη ε, γραμμή, αλλά δεν θέλω να προδικάσω και το τι θα ζητηθεί αύριο στο εργαστήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Στην ε, μελέτη σας από τον Ιούνιο είπατε ότι υπάρχει μια σειρά από κράτη-μέλη που ε, έχουν ήδη κάνει κάποιες εκτιμήσεις για την ε, κατάσταση των τραπεζικών του συντριμμάτων ως τότε. Πώς πάει η κατάσταση ως το τέλος της χρονιάς. Ναι, κάποια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει τα στοιχεία τους ε, για το ε, σχετικό χρονικό διάστημα. Το, ε, το χρονικό διάστημα καλύπτεται αλλά για κάποια ιδρύματα δεν έχουμε ακόμα όλα τα στοιχεία. Πρέπει κάποιοι να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους, ε, κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση στις χρηματαγορές. Θα χρειαστούν λοιπόν ε, και άλλα στοιχεία. Δεν έχουμε λάβει νέες αποφάσεις από το καλοκαίρι. Οι αποφάσεις τις οποίες τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία να λάβουμε είναι δευτερογενείς. Ελπίζω όμως ότι η σφαιρική εικόνα ε, έχει σχεδόν συμπληρωθεί. Δεν λείπουν πολλά κομμάτια του παζλ. Αλλά για το σύνολο της μεταβατικής περίοδου θα χρειαστούμε και άλλο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Και κινούμε και σε μια άλλη κατεύθυνση και μπορώ να το πω και εδώ δημοσίω. Έχουμε δύο πυλώνες για να μπορέσει μια τράπεζα να διασωθεί, να εξηγενθεί. Ετήσιο το ένα σύστημα και το άλλο η πρόσβαση στο FMI, δηλαδή η συνέχεια των ε, επιχειρήσεων και των συναλλαγών. Κάποιες από τις τράπεζες αυτές τις έχω πλησιάσει, έχουμε συζητήσει και έχω πει, εάν έχετε ε, μια σοβαρή ε, δυσκολία στον ένα πυλώνα, ο άλλος μπορεί να σας βοηθήσει να τα πάτε καλά. Ε, ο συνδυασμός και των δύο δηλαδή μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να μείνουμε ρεαλιστές και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Λαλιούκ από τους Σοσιαλιστές, η κυρία Λαλιούκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που έρχεστε συστηματικά για να μας ε, ενημερώσετε για τη δουλειά σας και τις εξελίξεις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά για μας. Και έρχομαι και εγώ ε, με συνάχη. Ελπίζω ότι αυτό που του μασουλάω θα με βοηθήσει να μην φταρνιστώ και να σας μολύνω με τα μικροβιά μου. Τώρα για τις κλιματικές αλλαγές πρόσφατα είδαμε το τι γίνεται με την παρουσία των, ε, δευτερογενών, των παραγόγων προϊόντων και το τι γίνεται και με τα trade books. Ε, είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πουληθούν, να τα ξεφορτωθεί κανείς και η υπόθεση δεξιά σέρνεται ακόμα. Ήθελα λοιπόν την άποψή σας για το θέμα αυτό και κυρίως για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα παράγωγα, ιδίως στην περίπτωση των trading booths ε, είναι σημαντικό να δούμε τι ρόλο μπορούν να αναλάβουν οι ρυθμιστές ε, και αν το προϊόν αυτό μπορεί να το χειριστεί κανείς. Η σχολή του Σικάγο είναι ελεύθερη. Αυτό που προτείνουν η αδειοδότηση για τη θέση σε εμπορία κάποιων χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι μια λύση. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση. Βλέπουμε κάθε μέρα να έρχονται μελέτε επιμελετών για του ε, οικονομικού κινδύνου και τι απειλέ και σε σχέση με τι κλιματικέ αλλαγέ από χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Εσεί πώ θα ενσωματώσετε το θέμα των περιβαλλοντικών απειλών και κινδύνων στη δουλειά σα και μετά δεδομένου του δικτύου κεντρικών τραπεζών και των, των, ε, των προέδρων τους για, την, ε, ε, για τον υπολογισμό του ε, κινδύνου. Ήθελα να ρωτήσω εάν το Συμβούλιο σας συμμετέχει και εάν είναι κάτι που το σκέφτεστε και το έχετε υπόψη σας και σκοπό να το αναλάβετε στο μέλλον. Να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά. Ας δούμε τι γίνεται με τα trading books και τα παράγωγα. Αυτό είναι σαφώς για μας προτεραιότητα. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω ε, λέγοντας ότι μπορούμε να δούμε τι είχε συμβεί με τη χρηματοοικονομική κρίση ε, και πού φτάσαμε σήμερα. Ένας τομέας που ανησυχούσε πολύ ε, έχει αλλάξει, έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα, η κεντρική αντισυμβαλόμενη. Η πλειονότητα δεν γίνεται πλέον σε επίπεδο λιανικής, ε, εμπορικό, αλλά σε επίπεδο κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Και για τον συστημικό κίνδυνο το κοιτάζει και η Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε είναι να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα αυτά και τι κάνουμε με την αφαιρεγκαιότητα. Μια από τις δουλειές που έχουμε αναλάβει και το κοιτάζουμε ανά περίπτωση, κάποιες υποθέσεις τραπεζών, μεγάλα χαρτοφυλάκια συγκεκριμένα, τους ζητάμε να μας προτείνουν ε, συστήματα και τι γίνεται αν ε, κλείσει κάνουλα, αν μπορούν τα βιβλία τους να τα κρατήσουν ανοιχτά, τι ανάγκη θα έχουν για ρευστότητα, πόσο θα χρειαστούν για να κλείσουν τα βιβλία και ούτω καθεξής, διότι πάντοτε βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι με την εξυγίανση τη Δευτέρα ξεκινά κανείς την αδιάρθρωση και μετά αρχίζει να βλέπει τα θέματα ένα προς ένα. Οπότε τεχνική δουλειά είναι ουσιαστικά η ανάλυση των λεπτομεριών ε, για την αφαιρεγκαιότητα προκειμένου να φτάσει κανείς στην πτώχευση τέλο πάντων σε κάτι ανάλογο. Το βασικό πρόβλημα είναι οι ανάγκες ρευστότητας που υπάρχουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν θα πήγαινα τόσο μακριά ώστε να πω ότι πρέπει κανείς να απαγορεύσει τα προϊόντα αυτά. Πρέπει όμως να κατανοούμε ποιε είναι οι σχέσεις που τους επιτρέπουν να λειτουργούν και πώς προχωρούν. Και επίσης κάτι που διαφέρει από την καθημερινή μας δουλειά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ομάδα κεντρικών τραπεζών, αυτό το δίκτυο και παρακολουθούμε λίγο από το περιθώριο από τα παρασκήνια. Δεν είμαστε μέλος του δικτύου κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι η κλιματική κίνδυνη, οι κλιματικές απειλές προς στιγμήν για μας θα έπρεπε να πάνε στα χέρια των εποπτών παρά στις αρχές εξυγίανσης. Πάντως, είναι ένα θέμα που και αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε στενά. Thank you very much. Now, Luis Ευχαριστούμε. Από το Ρινιό, ο κύριος Γαρικάνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που αναφέρατε για την σημασία της ρευτότητα και της εξυγένσης και για όλα αυτά που χρειάζονται. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα όμως στο πεδίο των δικών σας αναρμοδιοτήτων να μου πείτε πώς ε, βλέπετε να λειτουργεί το πλαίσιο για την εξυγίαση. Μήπως θεωρείτε ότι το κατόφλι έχει οριστεί υπό υψηλά και αυτό θα οδηγήσει στο να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ο ενιαίος μηχανισμός εξυγένσης. Υπάρχουν ήδη Ιταλικές τράπεζες οι οποίες ε, δημιουργήσαν προβλήματα, μιλώ για την τράπεζα του Βένετο και το ενιαίο ε, το, το Συμβούλιο εξυγένσης θεώρησε ότι δεν τηρούσαν τους κανόνες. Έχουμε επίσης ε, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η οποία το 2018 δήλωσε 2,7 δισεκατομμύρια ζημίες και δεν φαίνεται η ανακεφαλαιοποίηση να ξεπερνάει τα προβλήματα και να ε, αποδεικνύει τον, την ε, αξία της στην αγορά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, δημιουργείται η εικόνα ότι αυτό το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες αυτές να επωφελούνται δια των εκεφαλαιοποίησεων από λεφτά των φορολογουμένων. Είναι κάτι ξεκάθαρο στην περίπτωση της τράπεζας της Αξονία και, στην, και για τις Ιταλικές. Επομένως, τι θα κάνουμε για να σταματήσουμε κάποιες τράπεζες να ε, χρησιμοποιούν το σύστημα έτσι ώστε ουσιαστικά να μας αναγκάζουν να κάνουμε ό,τι θέλουν και να αποφεύγουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Απάντηση. Κατά την άποψή μου το κατόφλι δεν είναι υπερβολικά υψηλό. Γνωρίζω βέβαια όλο το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την διαφορά μεταξύ εξυγίανσης και πτώχευσης. Φέτος δημοσιοποιήσαμε ένα έγγραφο με το οποίο περιγράφουμε πώς θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία για την, για την αξιολόγηση του κατά πόσο μια τράπεζα εμπέπτει στο δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, εάν θα επιδιώξουμε μια εξυγίανση ή αν θα επιδιωχθεί μια ε, συντεταγμένη εκαθάριση. Μπορεί κανείς αυτό να το εφαρμόσει πιο αυστηρά, μπορεί να το αφαιρώσει με, με, με λιγότερη μεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερο αυστηρά. Ε, ωστόσο φοβάμαι ότι αυτός που, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι επειδή δεν γνωρίζουμε πώς θα λειτουργούσε μια καθάριση, να επιλέγουμε να πάμε στη λύση της εξυγίανσης. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια συζήτηση για το πώς θα λειτουργεί η ίδια η εκαθάριση, η συντεταγμένη εκαθάριση. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει και μια ουσιαστικότερη συζήτηση, μήπως θέλουμε περισσότερες τράπεζες να οδηγηθούν στην εκαθάριση, αν ε, συγγνώμη, στην εξυγίανση και αν ναι θα χρειαστεί να αυξηθούν και αντίστοιχοι πόροι των ταμείων ή αν όχι να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία για την εκαθάριση και για το πώς θα τις αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν προσπαθώ να κάνω κάποιο σχόλιο που να αναφέρεται σε συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής θα ήταν δίκαιο να πει κανείς ότι ο μηχανισμός της εξυγίανσης έχει λειτουργήσει, όμως όταν πάμε σε καθάριση, δεν είναι ξεκάθαρο ποια εργαλεία το χρησιμοποιεί κανείς. Και ανάλογα με την ισορροπία που θα επιλέξει κανείς θα πρέπει να ενισχύσει και τα αντίστοιχα εργαλεία του. Κύριος Γαρικάνο, η αλήθεια είναι όμως ότι αν ήμασταν περισσότερο γενναιόδοροι με το σύστημα εξυγίανσης, θα είχαμε λιγότερα προβλήματα με τα ενδεχόμενα να χρειαστούν εγκαθαρίσει. Καταλαβαίνω τι λέτε και καταλαβαίνω πω δεν θέλετε να μπείτε στι εθνικέ ε, σε εθνικά ζητήματα, αλλά απάντηση. Ναι και όχι. Ε, θα μπορούσε μια μεγαλύτερη γενοδορία στο Ταμείο για την Εξυγίαση να λύσει κάποια προβλήματα, όμω μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλε συζητήσει, όπω για παράδειγμα τα ελάχιστα κεφάλαια. Απαιτείται μια συγκεκριμένη κεφαλαϊκή επάρκεια από τι τράπεζε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η εκαθάριση ίσως να είναι μια καλύτερη λύση. Ε, ε, θα, θα, θα, θα πρέπει κανείς μάλλον να είναι προσεκτικός να μην δοθεί εντύπωση ότι η εκαθάριση είναι μια καλύτερη λύση γιατί ίσως αυτό οδηγήσει σε περισσότερες εκαθαρίσεις χωρίς να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει το ουσιαστικό πρόβλημα, το δομικό. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα της επικοινωνίας των τραπεζών με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και ε, όπως έχω πει και στο παρελθόν αυτή θα πρέπει να ε, ταιριάξει και με το πλαίσιο για την ε, καθάριση και με το πλαίσιο για την εξυγίαση. Από τους Πρασίνους, ο κύριος Ακελουγιονασέ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κιόνιξ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και για την συζήτησή σας μαζί μας. Αναφερθήκατε εκτενώς στα MRL, στις κεφαλαιακές απαιτήσει ε, είναι σημαντικό ε, ο τραπεζικός τομέας να κλείσει το κενό ε, της αναντιστοιχίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι προχωράτε με το θέμα αυτό. Μία επίκριση όμως παραμένει ότι δεν είναι ανοιχτός και διαφανής ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται στα ε, εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσει ε, στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναλογία. Πότε πιστεύετε ότι θα ανοίξουν τους λογαριασμούς τους και θα μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσει τους και έτσι και για την φερεγγιότητά τους και τη δυνατότητα εξυγίανσης. Μιλάμε για κεφάλαια διάσωσης ε, ε, και για κεφάλαιο ε, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Πότε πιστεύετε λοιπόν ότι θα κλείσει το κενό αυτό και πότε θα είναι διαθέσιμα σε όλους μας οι πληροφορίες αυτές. Τι είχαμε την συζήτηση αυτή ήδη στο PRRD1 και είχαμε πει ήδη από την αρχή ε, και είπαμε ότι δεν υπάρχει ε, υποχρέωση και έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ε, τα MRL. Είναι πολύ πλοκός ο υπολογισμός αυτός. Πάντα καλούσαμε όμως τις τράπεζες να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να είναι διαφανής όσον αφορά το παθητικό τους, ώστε να ε, αν επενδύσει κανεί να γνωρίζει πού ακριβώ βρίσκεται στι επενδύσεις αυτές. Ε, και δεύτερον, ε, είπαμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση να δημοσιεύουν οι τράπεζες τα στοιχεία των ελάχιστων απαιτήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι βλέπουμε ότι ε, αρκετές τράπεζες δημοσιεύουν τα νούμερα, ε, βέβαια κυρίως οι τράπεζες ε, όπου όλα είναι καλά. Βλέπουμε όμως αρκετές ε, τράπεζες και από τις άλλες να δημοσιεύουν ε, τις ελάχιστες απαιτήσει. Δεν βλέπω όμως να δίνεται πολύ προσοχή στο θέμα αυτό από τα μέσα μαζική ενημέρωση. πιο πολύ επικεντρώνονται σε άλλα στοιχεία. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και με ε, τον ΕΣΜΑ, την ε, αρχή της εσωτερικής αγοράς ε, και έχουμε αφήσει τον ΕΣΜΑ να αποφασίσει αν θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο θέμα αυτό. Πάντως είναι ένα γενικό θέμα που ισχύει και για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης μιας τράπεζας. Το 2022-2023 ε, σχολιάζουν οι Βρετανοί φίλοι μας να το σχολιάσουν αυτό, αλλά για μας είναι σαφές ότι το BRD και το SMA δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Ε, και πάλι αναρωτιέμαι πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά ναι, είναι ένα θέμα που πρέπει να, εξετάσουμε και ενδεχομένως να πρέπει να ε, σκεφτεί και ο νομοθέτης. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Φρανσίσκα Ντονέρτο από το ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω Ιταλικά. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα συμφωνήσω με την ερώτηση που μόλις έθεσε ο συνάδελφος για τα θέματα διαφάνειας. Διότι, όπως γνωρίζουμε, ο τρόπος που λειτουργεί ο ενέργειος μηχανισμός εξυγένσης καθώς και αυτός της ενιαίας αποπτίας ε, ακολουθούν πολύ περίπλοκες διαδικασίες. Γι' αυτό το πώς συνανούνται με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρώπης αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο πολλές φορές δεν είναι αρκετά διαφανές. Ε, διαφανής. Ε, τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις, που γίνονται οι ταξινομήσεις και κατηγοριοποιήσεις και το που βασίζεστε, σε τι δεδομένα, δεν ε, διατίθενται στην γνώση των υπευθύνων ούτε καν των βουλευτών. Και λέτε ότι η δημοσιοποίηση θα ήταν κακή για τι χρηματαγορέ και τον τρόπο που λειτουργούν. Όμω, για λόγου λογοδοσία και οι βουλευτέ και οι ελεγκτέ του ελεγκτικού συνεδρίου θα έπρεπε να έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες. Γνωρίζουμε καλά ότι τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται γίνονται υπό συνθήκες ιδιαίτερα, συνθήκες απορρίτου για να το πω έτσι. Εδώ λοιπόν μιλάμε για, μια, για ένα πλήγμα στη δημοκρατία και ακόμη ε, τα μενότατα στελέχη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, εντοπίζουν ότι είναι θέμα θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Ήδη στι 14 Ιανουαρίου του περασμένου έτου, το Ελεκτικό Συνεδρίο ζήτησε από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο να ακολουθούνται αυτοί οι κανόνε και για τι ανακοινώσει ε, που γίνονται προς το ελεκτικό συνέδριο εν γέννη και το Ευρωκοινοβούλιο στη δική σας περίπτωση. Εσείς τι θεωρείτε λοιπόν, θα έπρεπε αυτή η διαδικασία διαφάνειας να ισχύει για όλους, να δίδονται ακριβείς πληροφορίες στους άλλους θεσμικούς συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Εθνικές Βουλές, ώστε να μπορούν να, κάνουν αποφάσεις, να λάβουν αποφάσεις ε, τεκμηριωμένες. Και Εφόσον έτσι συμβαίνει, τι εργαλεία θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε. Νομίζω ότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή διαχωρισμού. Εδώ τα προγράμματα εξυγίανσης που βλέπουμε στην, ε, ε, ανάκτηση μάλλον που βλέπουμε στην, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολογούνται εκεί οι δικοί τους οι κοιτάζουν και ε, δίνουν την άποψή τους, ε, τις συμβουλές τους για οποιοδήποτε πρόγραμμα ε, διάσωσης ή εξυγίανσης. Αναφέρατε το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο αποτίμησε σε μια πρώτη έκθεση τον τρόπο που δουλεύουμε και ζήτησε τα προγράμματα εξυγένσης κάποιων θεσμών κάποιων ιδρυμάτων μάλλον. Αυτό μας ανησύχησε διότι τους επιτρέψαμε τα δουν υπό πολύ αυστηρά κριτήρια για τη δική μας την εξυγίανση. Ε, ο στόχος είναι τι θα κάναμε εάν. Εάν αυτές τις υποθέσεις τις δημοσιεύσει κανείς πολύ νωρίς, οι αγορές μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικά. Οπότε να μαντέψουν που θα πρέπει να προσανατολιστούν, διότι καταλαβαίνουν ποια είναι η βασική γραμμή συλλογισμού η δική μας και ξέρουν τι μέσα διαθέτουν, που ε, πιστεύουν ότι θα πρέπει να ε, δράσουν περισσότερο και πρέπει να είμαστε εδώ ιδιαίτερα επιφυλακτικοί προσπάθησα να το απαντήσω διαφορετικά. Είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε διαφανεί για τον τρόπο που χαράζουμε την πολιτική μα, τι προσδοκίε μα, αλλά όπω έχω πει και προηγουμένω, πρέπει να δούμε το αν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε περισσότερα για τα ε, αυτό δεν είναι πρόβλημα αλλά για την ε, Τράπεζα της Αγγλίας ή για τους Αμερικανούς συναδέλφους. Οι ίδιοι αξιολογούν την θερεγγιότητα και δημοσιεύουν κάτι στην Αγγλία. Στην, Αμερικα... στην Αμερική έχουν άλλο σύστημα. Πρέπει να δημοσιεύουν βασικά στοιχεία του τίτλου 1 και τα και τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και η Κεντρική Τράπεζα λέει ουσιαστικά αν είναι αρκετά ή μη αρκετά. Ε, μια βαθμολόγηση κάνω. Θα πρέπει να, εργαζόμαστε, να εργαστούμε από αυτού πολύ σκληρά. Το άρθρο 88 έχει αυστηρούς κανόνες περί απορρίτου για μας και ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ εύλογο αυτό. Οπότε πρέπει να πω ότι έχουμε ένα δεύτερο έλεγχο για τις επιδόσεις μας από το ελεγκτικό συνέδριο στα πέντε χρόνια λειτουργίας μας ως SRB. Οπότε είμαστε νομίζω παράλληλοι σε σχέση με το τι κάνει για το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα βρίσκω συσσωροποιημένα. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η κυρία Χιούμπνερ από το ΕΛΚ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις από εμένα. Η πρώτη έχει σχέση με το Brexit. Εάν σωστά ενθυμούμε, πριν από ένα χρόνο ή λίγο περισσότερο, λεγόταν ότι οι διάφορες τράπεζες θα μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατήσουν το διαβατήριο, την πρόσβασή τους στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Και ότι αυτό θα το έκαναν με τρόπο στρατηγικό, και το ερώτημά μου προ εσά είναι, θεωρείτε ότι αυτό απεφεύχθη ή εν πάση περιπτώσει πώ αξιολογείτε εσεί αυτό το φαινόμενο, θεωρείτε ότι συνέβη ή ότι καταφέραμε να το αποφύγουμε. Το δεύτερο μου ερώτημα έχει σχέση με την σχέση μεταξύ των αρχών ε, εξυγίαση και των αρχών εποπτείας. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να κάνουμε μια σύγκριση με αυτό που μας λέτε σήμερα σε σχέση με αυτό που μας έλεγε το θεσμικό όργανο που εκπροσωπείται όταν ξεκινούσε. Όσον αφορά τον καταμερισμό εργασίας, που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην αρχή της εποπτείας και την αρχή της εξυγίανσης. Με την εμπειρία που αποκτήσατε λοιπόν. Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει πραγματικά να αφορούν την αρχή εξυγίανσης και να μην τα παραπέμπει κανείς στην αρχή εποπτείας. Δεν μιλώ βεβαίω για το νομικό πλαίσιο, για τα θεσμικά που είναι ήδη δεδομένα, αλλά ποια είναι τα προβλήματα που εσείς πιστεύετε ότι στο θεσμικό επίπεδο ανήκουν στο δικό σας όργανο. Απάντηση. Σε σχέση με το Brexit και πράγματι τώρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στο Brexit στην πρωτολογία μου, να σας ενημερώσω ότι θεωρώ ότι έχουμε πολύ αποτελεσματικά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, καταφέρει να περάσουμε το μήνυμα προς τις ε, τράπεζες ότι θα χρειαστεί εάν δημιουργήσουν και αναλάβουν δραστηριότητες στην ε, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 27 κράτη-μέλη, ε, θα πρέπει να τηρούν τους αντίστοιχους κανόνες, να έχουν μια αντίστοιχη δομή ε, διοίκησης και κεφαλαϊκή επάρκεια. Εμείς καταφέραμε επίσης να συνεργαστούμε και με τις αρχές της αντίστοιχης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία. Ε, στόχος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι να συνεργαστεί με την αντίστοιχη αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ευρώπη για να δει εάν η τράπεζα είναι εξηγιάνσιμη στο κάθε μια από αυτά τα ε, περιβάλλοντα. Πιστεύω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε πρόοδο εδώ. Υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι έχουμε το, τις εκδόσεις ε, με βάση το αγγλικό δίκαιο. Ε, πολλές τράπεζες έλεγαν ότι πάντοτε εμείς έτσι ε, εκδίδαμε τα προϊόντα μας, αλλά φαίνεται ότι πολλές τράπεζες επιλέγουν είτε να ξεκινήσουν να κάνουν νέε εκδόσει εντό εκτός του πλαισίου των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε να δημιουργήσουν μια δυνατότητα, μια ασφαλιστική δικλίδα για να μπορούν να περάσουν σε αυτές τις εκδόσεις αν χρειαστεί. Για το δεύτερο σας ερώτημα. Πιστεύω ότι όταν ξεκινούσαμε στα πρώτα μας βήματα, συζητούσαμε πολύ την ανταλλαγή πληροφοριών και Πώ θα υπάρχει μια γενικότερη συνεργασία. Αυτό το κλείσαμε. Έχουμε πλέον ένα μνημόνιο συνεργασίας που ε, περιγράφει αναλυτικά πώς γίνεται και η ανταλλαγή πληροφοριών και οποτεδήποτε υπάρχει πρόβλημα θα έλεγα ότι το πρόβλημα έχει περισσότερο σχέση με τα πρόσωπα παρά με το σύστημα πια. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια καθημερινή συνεργασία και θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο ότι η εποπτική αρχή αρχίζει να, παρακολουθεί μια τράπεζα όταν ξεκινάει να έχει προβλήματα και προσπαθεί να την βοηθήσει να ανακάμψει, να αναδιαρθρωθεί, να βρει μια λύση. Ο στόχος τους είναι να βρουν μια λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα. Η δικιά μας οπτική γωνία είναι διαφορετική. Εμείς προσπαθούμε να εξετάσουμε, έχουμε φτάσει μήπως στο σημείο που πρέπει να πούμε ότι φτάνει πια και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια φυσική ένταση μεταξύ αυτών των δύο αρχών, η οποία είναι και απαραίτητη, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να δίνουμε την εντύπωση ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κινδυνεύει να καταρρεύσει υπερβολικά νωρί, αλλά ούτε και υπερβολικά αργά. Γιατί για να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, εάν κάποιος προσπαθήσει να, να διαρθρώσει έναν όμιλο, να τον βοηθήσει να ανακάμψει, πρέπει αυτός να έχει και μια αξία στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν να, τον, ε, να την έχει χάσει αυτή την αξία. Ε, επομένως θα έλεγα ότι μετά από αυτά τα χρόνια έχουμε βρει τη σωστή ισορροπία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλφρέτ Σάντες, σας ευχαριστώ πολύ. Όλο και περισσότερο η κατάσταση των μικρομεσαίων τραπεζών, πόσο μάλλον αυτών στα μικρότερα κράτη-μέλη, ε, αποτελεί ε, πηγή ανησυχίας. Ε, κάποιοι κατηγορούν τις ήπιε πολιτικές τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την κατάσταση αυτή, αλλά αυτό απέχει πολύ από την πλήρη εικόνα. Ε, προτάθηκε οι τράπεζες αυτές ε, να ε, μπουν σε καθεστώς παρακολούθησης. Έχουμε τα πρότυπα Βασιλείας 3 που έχουν σχεδιαστεί όμως για αμερικανικές τράπεζες. Ε, είναι ε, απαραίτητες οι ελάχιστες απαιτήσει, ε, αλλάζουν όμως συνεχώς. Και επίσης οι προσπάθειες ελέγχου των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν ενταθεί. Η κατάσταση λοιπόν ε, επιδεινώνεται συνεχώς. Κάποιοι διευθυντές τραπεζών ε, πιστεύουν ότι αποτελούν στόχο των συστημικών τραπεζών ε, που θέλουν να τις εξαγοράσουν. Ωστόσο, πολλές από τις μικρές τράπεζες εξυπηρετούν μικρές αγορές ε, που δεν ενδιαφέρουν ε, τις μεγάλες τράπεζες. Ε, δεν θα πρέπει αυτό να το εξετάσει το, Ευρωπαϊκό, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Εάν όχι, γιατί όχι. Εάν ναι, ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. Πολύ θα ήθελα να είχα μαγικό ραβδί. Νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι η λύση όσον αφορά τις μικρομεσαίες τράπεζες είναι να ασχοληθούν με ε, διάφορα ρυθμιστικά μέτρα. Όπως είπατε όμως, ε, εν μέρη αυτό δικαιολογείται. Από την άλλη, ε, αν μία τράπεζα εξυπηρετεί μία τοπική μικρή αγορά, τότε σημαντικό είναι να διατηρήσει και την κερδοφορία της στην αγορά αυτή. Σχεδόν όλες αυτές οι τράπεζες Ε, θα ε, βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Εξυγίανσης ε, και όχι το Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές αρχές ώστε να μπορεί να γίνει σωστός σχεδιασμός της εξυγίανσης σε χώρες όπου υπάρχουν πολλές τέτοιες τράπεζες, να μπορεί κανείς να ακολουθήσει μία προσέγγιση ε, ώστε ε, αν μια από αυτές τις τράπεζες ε, χρεοκοπήσει να έχουμε αφαιρεγγιότητα στο πλαίσιο ενός εθνικού ή στο μέλλον ακόμα και ευρωπαϊκού συστήματος. Δεν έχω κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και το εξή. Οι τράπεζε θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα των ε, ε, ενεργειών τους, ε, θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες αγορές και κατόπιν να δούμε εάν πρέπει να συγκεντρώσουν κεφάλαια, θα πρέπει να αναπτύσσονται όσο τους επιτρέπει το κεφάλαιο τους. Δεν έχω πραγματική απάντηση να σας δώσω, όπως είπα, δεν έχω μαγικό ραβδί. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό είναι πρόβλημα για ανθρώπους ε, κοινωνικά, διότι συχνά ε, εξυπηρετούν κοινωνικούς ε, σκοπούς οι τράπεζες αυτές και τις αφήνουμε μόνες και έρημες. Η Ευρώπη ε, έχει πολλές και διαφορετικές ε, τράπεζες. Ε, ξέχασα όμως να αναφέρω ένα πράγμα, ότι εμείς δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ενοποίηση της αγοράς. Αντιδρούμε όταν υπάρχει αφαιρεγγιότητα. Δεν θέλουμε συγχωνεύσεις για να έχουμε μεγαλύτερες τράπεζες. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ωραία, ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, Καρολάιν και αλλά από το Ρινιού. Ευχαριστούμε κυρία Κένη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ ήθελα λίγο να δούμε το θέμα του χάσματος ρευστότητας. Φέτος αποφασίστηκε το Συμβουλίο να μην έχει πρόσβαση μόνο στο Ταμείο Ενιαίας ε, Διάσωσης, αλλά και στο Backstop. Είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αυτός πλέον και είναι μια πολύ καλή εξέλιξη γιατί υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερους πόρους σε περίπτωση μια σοβαρής οικονομικής κρίσης. Όμως η Banco Popular, η περίπτωση της έδειξε ότι μπορεί να πτωχεύσει μια τράπεζα λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Έκτοτε το πρόβλημα της ρευστότητα συζητιέται σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με την ε, φραγιότητα. Γι' αυτό λοιπόν με απασχολεί η άποψή σας για τη σχέση ρευστότητας και διάσωσης. Κάποιες φορές υπάρχουν τράπεζες που δεν μπορούν να καλύψουν κινδύνους ρευστότητα για κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το SRF ελπίζει, ε, ε, υποθέτουμε ότι είναι 65 δις. Και εγώ δεν θα ήμουν υπέρ του να είναι μεγαλύτερο το ποσό αυτό. Γιατί λοιπόν να μην παραμείνει εθνικός ο ρόλος της εξυγίανσης και διάσωσης. Νομίζω ότι ήδη θίξατε το θέμα του backstop. Αυτή τη συζήτηση ελπίζουμε να μπορέσουμε να τη θέσουμε επιτάπητο στις ερχόμενες εβδομάδες και αυτό θα είναι μια σαφής προτεραιότητα για μένα και για όλους τους συναδέλφους το backstop θα είναι και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα λογικό αντίστοιχο με το μέγεθος των πόρων μας δηλαδή το backstop στην ουσία είναι ένα δάνειο μια πίστοση που εμείς θα πάρουμε ως Συμβούλιο και θα πρέπει να αποπληρώσουμε εκθέτοντας ε, τις ε, συνεισφορές των τραπεζικών ιδρυμάτων η συζήτηση νομίζω ότι έχει λήξει ως προς την ρευστότητα και την εξηγένση ε, και από τον Banco Popular και πριν είχαμε υπόψη ότι την περίπτωση της, της πτώχευσης μια τράπεζας πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πως αρχικός λόγος είναι η έλλειψη ρευστότητας αλλά αυτό ε, πρέπει να το δούμε συνδυαστικά δηλαδή το επόμενο πρωί οι αγορές δεν θα θέλουν αμέσως να ασχοληθούν με ε, ένα ίδρυμα το οποίο διασώσαμε, ακόμη και αν είναι ασφαλέστερο, καλύτερα κεφαλοποιημένο και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη Παρασκευή, αν είναι Δευτέρα πρωί ή πρώτη μέρα. Αλλά χρειάζεται κάποιο είδους δάνειο, τελευταίο καταφυγείο για να το πω έτσι για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η διάσωση πάντως τέτοιων ετοιμάτων μπορεί να χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτηθεί μόνο από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος, της ευρωζώνης δηλαδή. Και η συζήτηση αυτή συνεχίζεται, αλλά για μένα αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι όταν κοιτάζουμε τον κίνδυνο που είναι εμφυής στην δανειοδότηση από πλευράς μας, δανειοδότηση ρευστότητας, ο κίνδυνο είναι περιορισμένο, διότι μιλάμε για τράπεζα σε διαδικασία εξυγίανση, διάσωση, ε, που έχει ανακεφαλοποιηθεί. Δεν θα έπρεπε να είναι σοβαρό ο κίνδυνο. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα που κοιτάζουμε και έχουμε διερευνήσει αλλά προς στιγμήν δεν είχαμε δει να υπάρχει φοβερή διάθεση να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαι βεβαία ότι εάν το χρειαστούμε θα το βρούμε και θα είναι μια λύση, διότι αν δεν έχουμε μια λύση για τη ρευστότητα την μέρα που θα χρειαστεί, δεν έχουμε και διάσωση. Ευχαριστούμε Έχουμε ακόμα μία ερώτηση από τον Πέδρο Μαρκέ. Ε, με συγχωρείτε, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προφανώς, λόγω της συζήτηση για την Τραπεζική ε, Ένωση, έχω κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Κένιγκ. Ναι, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη διάθεση και ένας ρυθμός για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Γι' αυτό έχω μία ερώτηση για το μηχανισμό ασφάλισης των καταθέσεων, το σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων, για τις ε, κρατικές τράπεζες, πόσο μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία με βιοποίηση. Εάν θέλουμε να ε, αλλάξουμε την διασύνδεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναλόγως με το τι ασφάλιση θα αποφασίσουμε και τι εξαιρέσεις. Και δεύτερον, αυτό που διευθετήθηκε κάποιος τους ε, έφερε σε άβολη κατάσταση, ιδίως κάποιους εκλογικές ε, περιφέρειες. Με το backstop λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα το δεχτούν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πείτε το σε αυτή την ακρόαση γιατί υπάρχει αυτό το επιπλέον backstop, αυτός ο μηχανισμός πέραν του SRF και για το πώς θα δούμε τις, τους τραπεζικούς ομίλους, τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους και το πώς χρησιμοποιούν το κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους. Εάν υπάρχει πλήρης ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων στις διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται τα τραπεζικά ιδρύματα, τι θα γίνει με τους μεγάλους ομίλους και πώς θα είναι λιγότερο διασώσιμα υποκείμενα σε εξυγίανση τι θα ισχύει η ρευστότητα και το κατά πόσον έχουν ρευστότητα αυτοί και οι θεατρικέ τους, τα ιδρύματα που εξαρτώνται από αυτούς. Ναι, να προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση, μάλλον στη δεύτερη ερώτηση πρώτη, διότι η πρώτη και η τρίτη κάπως ε, συσχετίζονται. Για μένα ο μηχανισμός του backstop ήταν 65 δις, αλλά εν τέλει είναι ένα ποσό το οποίο ελπίζουμε να μην χρησιμοποιήσουμε, αλλά είναι η έσχατη λύση εφόσον χρειάζεται κάποια στιγμή μια διάσωση. Και είναι περισσότερο για να καθησυχάσουμε τις αγορές και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να αντιδράσουμε αμέσως όταν χρειαστούμε τον backstop και να μπορούμε να πούμε ότι αν γίνει κάτι και έχουμε ένα μεγάλο ε, κλειδονισμό ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και να διασώσουμε το σύστημα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό βέβαια, τόσο πιο αξιόπιστο είναι και λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιηθεί. Η δεύτερη ερώτησή σα. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει αναβιοποίηση στο σύστημα ασφάλιση των καταθέσεων. Είπα ότι έχουμε κάποια συστήματα παράλληλα αλλά λίγο αντικρώμενα μεταξύ τους. Έχουμε την ευρωπαϊκή εποπτεία, έχουμε την ευρωπαϊκή εξυγένση και τα δύο λειτουργούν καταρχήν παράλληλα και όταν ε, δει κανείς τι γίνεται στην ομάδα όλων αυτών, ε, το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τη θηγατρική σε μια χώρα που μπορεί να πλήττει το εθνικό σύστημα καταθέσεων. Ε, τι, αυτό το χρησιμοποιούν κάποιο επιχείρημα για να πούν ότι χρειάζονται άλλες εγγύσεις, άλλες διασφαλίσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε τα εσωτερικά εμελεκτός των προσθέτων που θα απαιτηθούν και το ερώτημα που τελικά προκύπτει είναι ότι ένας όμιλος, ένα ίδρυμα μπορεί να μην είναι περισσότερο διασώ... διασώσιμος δυνατό να διασωθεί, να εξηγενθεί, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη κατανομή των διαφόρων προβλημάτων σε όλη την έκταση του ομίλου. Και για το άλλο πρόβλημα, δεν το ανέφερα εγώ αυτό, το συζητάνε όλες οι τράπεζες, αλλά πρώτα απ' όλα το είδαμε στον κύκλο του 18-19 και είναι μια βασική προτεραιότητα για το 2020 σαφώς. Πρέπει να ε, δούμε τους κανόνες του bail-in, τα λεγόμενα playbooks. Τι θα κάνουν οι τράπεζες τώρα σε περίπτωση του bail-in. Θα πρέπει να καταγράψουν ε, τα αξιόγραφα, θα πρέπει να καταγράψουν όλα τα στοιχεία, να γράψουμε όλα τα στοιχεία του παθητικού και οι τράπεζες να μας πούν κατά λεπτός πώς θα είναι προετοιμασμένες και πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά αν χρειαστεί. Ποια θα είναι τα τεχνικά βήματα που θα ακολουθηθούν. Διότι εδώ δεν είμαστε στις ΗΠΑ που υπάρχει ένα σύστημα για όλους, που είναι ενιαίο. Είμαστε στην Ευρώπη που υπάρχουν 19, 19 διαφορετικά εταιρικά δίκαια, διαφορετικές διαδικασίες και κανόνες για την πτώχευση. Οπότε οι τράπεζες θα πρέπει να το κάνουν αυτό και σε επίπεδο μετοχής εταιρεία και σε επίπεδο θηγατρικών και είναι πολύ εύκολο να πει κανεί ότι τις απώλειες τις στέλνει στη μετρική και στις θηγατρικέ στέλνει το κεφάλαιο, αλλά αν πρέπει να λειτουργήσει διασυνοριακά, τι θα γίνει εάν πρέπει κάπως να συμμαζευτούν, να συρρυκνωθούν για να διασώσουν την κατάσταση. Επίσης, πώς διασφαλίζουμε τις θηγατρικέ. και για να απαντήσω και σε εσά με κάποιο τρόπο. Ο κατακαιρματισμό του κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάποιε αλλαγέ στην κατανομή πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τι προσπαθίε μα. Ωραία. Ε, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέλη και όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε κυρία Κέρνιγκ. Οπότε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ξαναρχίσουμε στις 4.00 με το επόμενο σημείο στην εμείς διάταξη.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 So, uh, let's resume the meeting. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Σημείο 14 συν 15. Απαιτήσει για τις ε, πληρωμές των φορέων στην αγορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες για τις ε, πολύτιμες συνεισφορές τους στην συζήτησή μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής Αίκων για όλη υποστήριξη, για τις συμβουλές τους. Ήταν ε, πολύ σημαντικές για την ολοκλήρωση αυτής της κοινή δουλειά. Μιλάμε για διαδικασία διαβούλευσης και τις δύο εκθέσεις. Πρέπει να συντάξουμε ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για τις δύο προτάσεις. Πρώτος μου στόχος ε, με τις ε, εκθέσεις αυτές ήταν να λάβω υπόψη πέντε βασικές μέρημνες. Πρώτα απ' όλα την ψηφιοποίηση, μετά τη συνεργασία και την αναρμόνιση, τα think tank και τις τεχνολογίες στοιχειών, καθώς και την απλούστευση μας με την τεχνολογία. Καταλαβαίνω την διαδικασία διαβούλευσης, το Συμβούλιο έχει ήδη φτάσει σε συμβαστική λύση για το τελικό κείμενο, Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να επαναλάβουμε την δέσμευσή μας να εργαστούμε το του θέματος. Οι απάτες ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικές για τις εθνικές αρχές και η ηλεκτρονική επικοινωνία ε, διωγγώνει με τις διασυνοριακές συναλλαγές το μέγεθος του ΦΠΑ και της απάτης του. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται ετησίω και η απάτη γίνεται όλο ένα και πιο εξελιγμένη και απαιτεί και τέτοιες προηγμένες αποκρίσεις από τους συνομοθέτες και τις διοικητικές αρχές. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο αποφάσισα να μην χρησιμοποιήσουμε απλουστευμένη διαδικασία, με ένα μοντέλο στην εποχή, κατάλληλο για την εποχή της ψηφιοποίησης και να γίνει αυτό μια κορυφαία προτεραιότητα. Θέλουμε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το θέμα το Δεκέμβριο και επευκαιρίες να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και την υποστήριξη για το αίτημα της ομάδας μου να περιληφθεί στην ατζέντα της Ολομέλειας το σημείο. Και για τον κανονισμό και για την οδηγία, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα για τον κανονισμό. Είχαμε 23 τροπολογίε που υποβλήθηκαν. Πηγαίνουν όλε στην ίδια κατεύθυνση. Περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, λεπτομερή δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, περισσότερε συμβαστικέ λύσει από τα κράτη-μέλη και ένα ενισχυμένο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι οι προτινόμενε συμβαστικέ λύσει είναι καλά εξισορροπημένε, αναφέρουν σωστά τι προτεραιότητέ μα να υπάρχουν ίσοι κανόνε ανταγωνισμού για τη διοικητική συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών για την οδηγία. Έχουμε 45 τροπολογίε. Οι περισσότερε βελτιώνουν το σύστημα υποβολή εκθέσεων, συμπληρώνουν την πρόταση, ε, όπω και οι τροπολογίε ε, επί του κανονισμού που μόλι ε, τι σχολίασα και νομίζω ότι το Συμβούλιο έχει μια θέση ικανοποιητική με την διαδικασία της διαβούλευσης, έχει έτσι και τον τελευταίο λόγο σε κάθε περίπτωση εμείς μπορούμε να εντοπίσουμε τις δικές μας προτεραιότητες και τις εναλλακτικέ απόψεις. Οι, ε, διαφορές, οι διαστάσεις απόψεων προκύπτουν για τις απαιτήσει ε, πληρωμών ε, είναι σαφή στη συζήτηση αυτή. Από την πλευρά μου πιστεύω ότι μπορούμε να εξισορροπήσουμε την θέση του Συμβουλίου με τις δικές μας απόψεις, με περισσότερες φιλοδοξίες και τις προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον. Έχουμε διαφορετικές προοπτικές για τα δύο σημεία και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται ε, για τους παρόχους ε, υπηρεσιών πληρωμών ε, είναι ένα από τα θέματα αυτά, αλλά έχω αισιόδοξη στάση. Μπορούμε να βρούμε εξορροπημένες προτάσεις και για, τις δύο, και για τα δύο σημεία με σωστή προτεραιότητα για να βρούμε τα μέτρα που θα καταπολεμήσουν πράγματι την απάτη ΦΠΑ και να συμβάλλουμε στι γενικέ προσπάθειε να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία για φορολογικά θέματα. Πιστεύω ότι σήμερα έχουμε ευνοϊκέ προποθέσει για να εγκρίνουμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου που να είναι πιο φιλόδοξη από αυτή του Συμβουλίου. Αν το κάνουμε αυτό, λέμε ότι θέλουμε περισσότερη συνεργασία αλλά και περισσότερη αφοσίωση στην καταπολέμηση τη φορολογική απάτη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you now for, uh... Σας ευχαριστούμε. Κυρία Καρολίνα Ντερή. Ζάμπα Μόλναρ, μάλλον πρώτα, τους σκιώδες από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Μόλναρ. Ευχαριστώ. Η δασιονοριακή απάτη ΦΠΑ είναι ένας τομέας που ανθεί δυστυχώς. Έχουν μέχρι και δημιουργηθεί μέχρι και εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων. Στην Ουγγαρία ο ΦΠΑ, ο συνήθις συντελεστής ΦΠΑ είναι 20% που είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι ο υψηλότερος, και αυτός μας κάνει πόλο έλξη για τέτοιου τύπου απάτες ΦΠΑ. Έχουμε, έχουμε ε, ε, εταιρείε οι οποίες πέραν από την ειδικευσή του στον φορολογικό σχεδιασμό ειδικεύονται και στην απάτη ΦΠΑ. Βοηθούν επιχειρηματίε, ουσιαστικά να φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των τραπεζών και των αρχών όπως αναφέρεται και στην πρόταση αυτή, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει να δημιουργηθεί το μητρό συναλλαγών, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι, ε, ποιες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη ΦΠΑ. Δεν θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι το προσχέδιο έκθεσης που μας υποβάλλει είναι εξαιρετικό με τις συζητήσεις που είχαν μέχρι στιγμής έχουν απομείνει διαφωνίες μόνο σε πολύ λίγα τεχνικής φύσης ζητήματα και είμαι αισιόδοξο ότι στο τέλος θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την τροπολογία που ζητά οι νέοι κανονισμοί να αρχίσουν να εφαρμόζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών, για όλων μας, γιατί όλοι θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την απάτη. Σας ευχαριστούμε, Αντρέ Κοβάικ, για το Ρινιού. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Εξαιρετική δουλειά έχει κάνει. Αναφέρθηκε ότι τα δύο αυτά θέματα είναι σημαντικά για να ε, καταπολεμήσουμε την απάτη ΦΠΑ. Αποτελούν ε, σημαντικό βήμα. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που ανέφερε και ο εισηγητής. Ε, πόσο σημαντικές είναι οι εκθέσεις αυτές για να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι για την ψηφιακή εποχή. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση ώστε να φροντίσουμε οι κανόνες ΦΠΑ και στο μέλλον ε, να ε, αντιστοιχούν στους στόχους μας, σε την καταπολέμηση της απάτης δηλαδή. Όσον αφορά την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας, ε, συμφωνούμε απόλυτα με την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος στην τριετία, δηλαδή αντί για τη διετία. Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, σχετικά με ε, τους ε, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το κείμενο με βάση την θέση του Συμβουλίου. Τον Οκτώβριο το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση και στα δύο αυτά θέματα κάποιες παρατηρήσεις για, κάποιους, ε, για κάποια θέματα. Την ε, υποβολή εκθέσεων, ε, την υποβολή συνολικών εκθέσεων για να μειωθεί το διοικητικό άχθος και επίσης οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν έχουν πάντα όλες τις πληροφορίες στα χέρια του. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάτι που δεν γνωρίζουν. δεν θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία που δεν έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, ε, σκοπεύουμε να υποβάλουμε τροπολογίε ακολουθώντας τη λογική αυτή. Ε, συμφωνούμε και όσον αφορά το κατώτατο όριο για την ε, υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Τέλος, συμφωνούμε και με τις συγκεκριμένες διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης καρουσέλ. Υπάρχει γενική συμφωνία. Νομίζω όσον αφορά την γραμμή που θα ακολουθήσει η έκθεση του Συμβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια για τη συνεργασία και τις συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε σήμερα κατά την ψηφοφορία την θέση μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς από τους πρασίνους που να θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Από το ID. Ούτε. Eugene Ζήκα από το ECR. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέρφους για την ε, πολύ καλή και επικοδομητική προσέγγιση τους. Νομίζω ότι έχουμε συνένεση σε μεγάλο βαθμό. Η απάτη ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης αυτής. Από τότε που ε, η ΕΚΟΦΗΝ κατέληξε στη γενική προσέγγιση της ε, πριν ένα μήνα, δεν είδαμε ε, σημαντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το άρθρο 113 της ε, συνθήκης λέει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει ομόφωνα να υιοθετεί αποφάσεις για την εναρμόνιση της ε, φορολογίας μετά από διαβούλευση με το Εθνικό Κοινοβούλιο η ιστοσελίδα του Συμβουλίου ε, ενημέρωσε σχετικά με τη γενική προσέγγιση στις 8 ε, Νοεμβρίου, ε, θεωρώντας ότι θα υιοθετηθεί το κείμενο από το Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω συζήτηση μετά από την γλωσσική και νομική αναθεώρηση του κειμένου. Η δήλωση αυτή δεν αναφερόταν σε διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ συμφωνώ απολύτως με την αρχή της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 113 τη συνθήκη, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ όλες οι διατάξεις του άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στην διαδικασία διαβούλευση. Ίσως γι' αυτό λοιπόν να ενδείκνεται το Κοινοβούλιο να ε, μεταφέρει αυτή τη θέση και στο Συμβούλιο. Στόχος της διαβούλευσης είναι συμβουλευτικός η διαδικασία αυτή ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει πολύ καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Περέιρα ε, για την, ε, και για τα δύο σχέδια εκθέσεων και ακόμη περισσότερο για τα compromises, για τις συμβιβαστικέ προτάσεις που μας έστειλε, που ε, δείχνουν ότι κατέβαλε μια προσπάθεια να συμπεριλάβει και αρκετές από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους οικειώδεις ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων. Διαπιστώνω μια ευρεία συνένεση από τις πολιτικές ομάδες, γιατί όντως η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι μια πληγή κοστίζει στις εθνικές οικονομίες, κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοστίζει ιδιαίτερα στους πολίτες που είναι συνεπείς και έντιμοι ή τις επιχειρήσεις που είναι έντιμες και πληρώνουν με περισσότερους φόρους αυτό που με την απάτη γλιτώνουν όσοι χρησιμοποιούν πλάγια μέσα. Και με αυτή την έννοια η φορολογική απάτη δεν ζημιώνει μόνο τα δημόσια οικονομικά. Ζημιώνει και τον ε, υγιή ανταγωνισμό γιατί δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την φορολογική απάτη. Η ίδια η Επιτροπή υπολογίζει ότι το εισόδημα που χάνεται από την φοροαπάτη είναι τεράστιο, 137 δισεκατομμύρια ευρώ και αν δούμε και την ανάλυση ανακράτος μέλος, εκεί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην έκταση του φαινομένου. Σε αυτό που όλοι όμως συμφωνούμε είναι ότι για να το περιορίσουμε αυτό χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Δεν μπορεί κάθε κράτος μέλος μόνο του να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναρωτηθούμε κιόλα για ένα θέμα όχι τόσο τεχνοκρατικό, αλλά πολιτικό. Γιατί οι περισσότερες αποκαλύψεις για θέματα φορολογικής απάτης μέχρι τώρα έχουν γίνει από μερικές δεκάδες δημοσιογράφους που κάνουν investigating journalism ή κάποιους whistleblowers και δεν έχουμε καταφέρει οι ευρωπαϊκές αρχές, οι μηχανισμοί των κρατών μελών ή της Κομισιόν να ανακαλύπτουν αυτά τα σκάνδαλα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναρωτηθούμε υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής βούλησης ή μας λείπουν επαρκείς μηχανισμοί εναρμόνιση της νομοθεσίας να κλείνουμε τρύπες και παράθυρα που επιτρέπουν στην απάτη. Και γι' αυτό νομίζω ότι οφείλουμε, και το κάνει η έκθεση με τις προτάσεις της, να ενισχύσουμε τη διοικητική συνεργασία, την εναρμόνιση, την ανταλλαγή δεδομένων και των πρακτικών, να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες ακόμη πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να κάνω ε, ορισμένες πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ε, ριζοσπαστικοί και τολμηροί σε μερικά πράγματα. Να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την την πρόσβαση στα δεδομένα. Με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, πιστεύω ότι τα δεδομένα πρέπει να κρατιώνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώνεται ο σχετικός έλεγχος και να μην εξασφαλίζεται η απάτη. Το δεύτερο, χρειάζεται πιο, αυστηρές, πιο αυστηρή τιμωρία των εταιριών που χρησιμοποιούν τη φορολογική απάτη. Και επίσης νομίζω ότι τα θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ θα πρέπει να τα δούμε πιο οριζόντια για να καλύψουμε μέσα εναρμόνισης νομοθετικά και διοικητικά κενά, καθώς οι επιχειρήσεις στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπαρίου εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα αυτά τα κενά για να ε, κάνουν φορολογική απάτη. Με αυτό το πνεύμα θα κινηθούμε και στην ψηφοφορία σε λίγες ώρες. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρολίνα Ντρί από την Γενική Διεύθυνση Ταξούτ. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα. Ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης που καταδεικνύει πόσο σημαντική θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταπολέμηση της απάτης και της ε, φορολογικής απάτης ακόμα περισσότερο. Όπως ε, ήδη αναφέρθηκε, είναι ένα διαρκές πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε διαπιστώσει ότι αναφέρεται και στις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής, η οποία θα επιδιώξει σε δύο, σε δύο, να προχωρήσει σε δύο προσεγγίσεις και να βελτιώσει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και να βελτιώσει τους μηχανισμούς καταπολέμησης της απάτης. Ευχαριστούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση που βάλει σε σχέση με την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι οι τροπολογίες που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέονται με όλα τα δύσκολα ζητήματα. Αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση, στην ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία, να βελτιωθεί η πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες και δεδομένα. Η πρότασή μας προσπαθεί να καλύψει κάποια από αυτά τα κενά σε αυτούς τους τομείς. Τα κενά αυτά τα βρίσκουμε και στις τροπολογίες σας, επομένως φαίνεται ότι όλοι έχουμε την ίδια νοοτροπία εδώ. Καλωσορίζουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες, ακόμα και εκείνες που θεωρούμε ότι ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογή που είχε προτείνει η Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε να τις ε, συζητούμε ορισμένε από αυτές. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της Eurofisk, η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων που είναι ε, διαθέσιμα σε σχέση με την απάτη. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου των υπευθύνων των φορολογικών αρχών από τα 27 κράτη-μέλη, στην οποία συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι από κοινού και πώς μπορούν να συνεργαστούν για να τα λύσουν. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή, ε, στις 6 Δεκεμβρίου, οργανώνουμε ένα συνέδριο για το ζήτημα του ΦΠΑ και ε, των τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τις αναφορές που υπάρχουν και στην έκθεση του Κοινοβουλίου για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να έχουμε καλύτερη συλλογή δεδομένων, για να έχουμε καλύτερη καταπολέμηση της απάτης και πώς μας επηρεάζουν σε όλα αυτά οι τεχνολογίες blockchain. Υπάρχουν επίσης κάποιες, τεχνολογίες, κάποιες οι οποίες πιθανώς να αποδυναμώσουν την πρόταση. Για παράδειγμα, Αναφέρομαι στην τροπολογία η οποία λέει ότι θα πρέπει να παραδίδονται τα στοιχεία όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωτικά. Εάν ε, υπερβάλλει κανεί σε αυτό και τα στοιχεία που ε, είναι διαθέσιμα είναι υπερβολικά συγκεντρωτικά, ίσω να μην έχει πρόσβαση στι μεμονωμένε συναλλαγέ που θα του επιτρέψουν να διαπιστώσει αν υπήρχαν απάτε. Ε, σε γενικέ γραμμέ πάντω υποστηρίζουμε και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με εσά. Σα ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και για τις ε, συνεισφορές τους σε αυτή τη συζήτηση. Το βασικό ζητούμενο σε αυτή τη συζήτηση είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές για την καταπολέμηση της απάτης, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων και διοικητική συνεργασία, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την απάτη ΦΠΑ άμεσα θεωρώ ότι η υπερψήφιση με μεγάλη πλειοψηφία ε, στην Επιτροπή και αργότερα στην Ολομέλεια ευελπιστώ ότι θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι εδώ ακολουθούμε τη διαδικασία ε, σύμφωνη γνώμη, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα δώσει ένα μήνυμα προ την Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό ελπίζω λοιπόν να είναι το αποτέλεσμα, ε, ξεκινώντας από την σημερινή μας ψηφοφορία, συνεχίζοντας με την συζήτηση στην Ολομέλεια και φροντίζοντας το θέμα αυτό να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη του δημοσίου διαλόγου και στα θέματα που απασχολούν τις πολιτικές ομάδες και που θα τις απασχολούν τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι για τα θέματα αυτά, ε, για, αυτούς τους, για αυτές τις δύο εκθέσεις, οι ψηφοφορίες θα γίνουν στις 5. Ο κύριος Μαυρίδης δεν φαίνεται να έχει έρθει ακόμα. Μήπως υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα τον ε, αντικαταστήσει. Όχι, από ό,τι φαίνεται... Ε, στο, στην ημερήσια διάταξη είχε προγραμματιστεί αργότερα αυτό το θέμα, γι' αυτό ίσως να μην έχει έρθει ο κύριος Μαυρίδης. Κάνουμε διάλειμμα δύο λεπτών. let's Ας ξαναρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο 16 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ετήσια έκθεση για το 2018. Εισηγητή, ε, ο κύριο Μαυρίδη από του Σοσιαλιστές και Δημοκράτε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστήρηση και η αλήθεια είναι ότι δεν θα τα χρειαστώ αυτά τα πέντε λεπτά. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συζητούμε για την ετήσια έκθεση της το 2018. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους Συνολικά 203 τροπολογίες, προτάσεις τροπολογιών επιβλήθησαν. Το επόμενο στάδιο είναι οι συναντήσει των σκιωδών για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ. Ο στόχος μου, κύριε Πρόεδρε, είναι να έχω την ίδια προσέγγιση με αυτή που είχα μέχρι τώρα. Δηλαδή, την προσέγγιση που ακολούθησα στη σύνταξη του κειμένου και εξηγούμε. Θα προσπαθήσω να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισορροπία, να είναι χρήσιμε οι προτάσει μα, να είναι επικοδομητικέ, αλλά όπου χρειάζεται δεν θα αποφύγουμε και την άσκηση κριτική. Ιδιαίτερα εστιάζοντα στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πολιτικών της. Και πάλι βέβαια λέγοντας ότι θα προσπαθήσω να επιδιώξω συμβιβαστικέ λύσεις, ε, τη συμφωνία των συναδέλφων όσο το δυνατόν περισσότερο. Με αυτό το σκεπτικό θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στο κείμενο συμβιβασμού όλες τις ιδέες που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους και τα κύρια ε, θέματα που θα εξετάσουμε στις ε, συναντήσεις των σκιωδών Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να κάνω και για να σας αναφέρω μερικά από αυτά τα θέματα είναι το εξή. ο αντίκτυπος των ε, πολιτικών της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωζώνη, ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία και στους ρυθμούς ανάπτυξης, η μελλοντική νομισματική πολιτική, η ε, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πολλά άλλα δεν προτίθεμαι αυτή τη στιγμή και στο επίπεδο που βρίσκεται η συζήτηση να ξεκινήσουμε μια συζήτηση επί των λεπτομεριών. Βέβαια μπορώ να πω ήδη ότι όταν έχουμε τροπολογίες οι οποίες ε, έχουν ε, διστάμενες πολιτικές κατευθύνσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον ε, κοινό παρονομαστή και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε συμβιβαστικές λύσεις. Φαντάζομαι ότι στην πλεονάτωτά του το σώμα επιθυμεί να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη, να ενισχύσουμε το ευρώ. Επομένως, αυτό με καθιστά αισιόδοξο ότι στο τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει το σωστό μήνυμα και τι σωστέ προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό προσβλέπω στις επικοδομητικέ και ενδιαφέρουσε συζητήσει που θα έχω με του συναδέλφου, στις συναντήσει των σκιωδών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε τρία λεπτά για τον καθένα από τους σκιώδους εισηγητές. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ευρά από το, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Μαυρίδη, για την επικοδομητική του δουλειά Ευχαριστώ και τους συναδέλφους του ΕΛΚ και τον ε, συντονιστή μας, τον κύριο Φέρμπερ, για τις τροπολογίες και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τώρα. Η σειρά τροπολογιών που υποβάλαμε έχουν να κάνουν αυστηρό με την εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εγγυηθούμε την ποιότητα τη έκθεση και κυρίω επιμείναμε σε κάποια σημεία την ανεξαρτησία τη ΕΚΤ την, ε, τον πρωταρχικό στόχο της νομισματικής πολιτικής που επιδιώκει η ΕΚΤ, δηλαδή την σταθεροποίηση των τιμών. Επίσης, θυμήσαμε ότι η νομισματική πολιτική δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις απαραίτητες διεθνωτικές μεταρρυθμίσεις και δώσαμε έμφαση στην ανάγκη να ξανασχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα την νομισματική πολιτική, ιδίως το πρόγραμμα των ε, αγορών στοιχείων του ενεργητικού. Όσο για την ε, ε, χαμηλή αύξηση, έχουμε μιλήσει για τις δυσμενείς συνέπειε για τους αποταμιευτές και τις κατάθεσεις τους. Και πρέπει να ε, επαγρυπνούμε και για τα κρυπτονομίσματα, τη σταθερότητα σχετικά, καθώς και τη σημασία των ε, μεσοπρόθεσμων πληρωμών, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ σε, στο διεθνές προσκήνιο. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά για να βελτιώσουμε την κατανόηση των αποφάσεων τη ΕΚΤ από του πολίτε, να γίνουν όλα αυτά πιο εύληπτα. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει για τι συμβαστικέ ε, τροπολογίε και να φτάσουμε σε συμφωνία στα πλαίσια τη Επιτροπή μα, τουλάχιστον το Γενάρη του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οι Ρινιού δεν έχουν στείλει κάποιον ε, σκιώδη, οπότε περνάμε στον κύριο Γιάκον Γιούνας από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μαυρίδη για τη δουλειά του. Μας δώσατε ένα πλαίσιο για το πώς θα συνεχίσετε την εξέταση του θέματος. Πολύ χρήσιμο αυτό. Ε, για τις τροπολογίες και για τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει από χθε και που συνεχίζεται ε, χθε με την κυρία Λαγκάρτ, ε, πρέπει να πω ότι τα θέματα αυτά δικατοπρίζονται και στις τροπολογίες μας, όπως τα θέξαμε Τώρα, από την πλευρά των πρασίνων, και θα ήθελα να αναφέρω κάποιες από τις προτεραιότητές μας. Ήδη το ανέφερε η συνάδελφος, ε, τα κρυπτονομίσματα για κεντρικές τράπεζες ως στοιχεία του ενεργητικού είναι ένα στοιχείο σημαντικό, πρέπει να το εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια και δεν είμαστε η μόνη ομάδα που θέλει να μιλήσουμε για crypto assets και όχι για cryptocurrencies απλώς, όχι κρυπτονομίσματα, αλλά κρυφά στοιχεία του ενεργητικού. Και θα πρέπει να δούμε πώς ενισχύεται ο ρόλος τους και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές συμβαστικές και για αυτό το θέμα. Στηρίζουμε την, ε, το να συνδυάσουμε τις προσπάθειες της ΕΚΤ με άλλες κεντρικές τράπεζες και να διερευνήσουμε τις προοπτικέ που ανοίγονται, τι προκλήσεις ε, που θα έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας των χρηματοπροστατικών, ε, είναι σημαντικό να δούμε και τις κλιματικές αλλαγές προφανώς. Οπότε συνιστούμε να προβλεφθεί εδώ ένα ιδιαίτερο τμήμα στην έκθεση, γιατί η Ένωση έχει ήδη αναλάβει σοβαρέ δεσμεύσει για την επιδίωξη των κλιματικών στόχων. Το έχει συζητήσει και η ΕΚΤ. Μόλι την περασμένη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαίωσε την ε, αφοσίωσή του να ταρθεί σε αυτόν τον αγώνα ε, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται πιστεύουμε και στην έκθεση. Γι' αυτό προτείνουμε ένα ξεχωριστό τμήμα για το θέμα αυτό. Για την ΕΚΤ και την ε, νομισματική της πολιτική. Σημειώνουμε ότι κάποιες τροπολογίες πήγαν ε, λίγο παραπέρα από ό,τι χρειάζεται ως προς τις συνέπειες της ε, πολιτικής της ΕΚΤ. Πιστεύουμε ότι η πολιτική ως τώρα που δεν είναι πάντοτε συμβατική, είχε κάποιες αρνητικές, κάποιες δυσμενείς συνέπειες σίγουρα, αλλά δεν πάβει να έχει και θετικές. Και θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα επικοδομητικά μέτρα. Η κριτική που θα ασκούμε να είναι και αυτή επικοδομητική και έχουμε σκοπό να στηρίξουμε τον εισηγητή. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε βεβαίως ε, την ε, ΕΚΤ μόνο. Υπάρχει και ο τομέα ε, των ιδιωτικών τραπεζών και μετά η ουδετερότητα στην αγορά εδώ θα πρέπει να αυτό το χρόνο να θεωρηθεί και αυτή η διάσταση και δεν θα πρέπει να έχουμε προκαταλήψεις στις επενδύσεις και θα πρέπει οι επιχειρήσεις και εταιρείε να συνεχίσουν ε, να οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, όμως είμαστε ανοιχτοί για να το συζητήσουμε και αυτός προς την εποπτεία. Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε από κενού τη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσει το αρχιτεκτόνημα της ε, χρηματοδοτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μια εναρμόνιση και ο ε, τομέα χρειάζεται στήριξη για τις τραπεζικές αρχές, για τον τομέα των ασφαλιών, για το τι συμβαίνει με τους καταναλωτές. Όλα αυτά είναι πολύ κατακαιρματισμένα προς στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να αντλήσουμε έμπνευση και από το μοντέλο από το μοντέλο Twinks και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις σχετικές συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο. Ισότητα των φύλων. Δεν υπάρχει ακόμα η εκπροσώπηση των φύλων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίω στον τομέα των εποπτών και των σωμάτων των φορέων της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Αυτό λοιπόν για μας είναι μια προτεραιότητα ε, και ε, προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία και συνεννόηση. Ευχαριστώ. Εάν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κανείς από την ID, Οπότε, ο λόγο στον κύριο Φανόφερφελτ από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους άλλους ε, σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο θέμα αυτό. Κατά την συζήτηση του σχεδίου έκθεσης ε, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος Έπινγκ πήρε το λόγο ε, στο όνομά μου, διότι εμένα με πίεζε ο χρόνος. Έπρεπε παράλληλα να ε, λαμβάνονται αποφάσεις. Ε, έπρεπε να είμαι παρόν στον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό. Ο συνάδελφος Έπινγκ και εγώ θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης περιέχει πολλά πολύτιμα στοιχεία έχουμε χάσει την ευκαιρία σε κάποια θέματα ε, για επικοδομητικές επικρίσεις απέναντι στις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει συνολικά 34 τροπολογίες, δεν θα τις διατρέξω όλες, απλά θα αναφερθώ στα κύρια σημεία συνοψίζοντάς τα σε πέντε θέματα. Καταρχάς, αυτονομία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι υψίστης σημασίας και γι' αυτό δεν συνάδει με την επιθυμία να συμμετέχει σε πολιτικές εκστρατείες. Ε, αυτό ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι κάτι που θα πρέπει να αποφύγουμε. Δεύτερον, ε, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει μου φαίνεται ε, κάπως περίεργο το ότι θα πρέπει να ε, ε, επηρεάζει την νομισματική πολιτική. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώνονται. Πιστεύω ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι αυστήρη, ενώ σε περιόδους κρίσεων θα πρέπει να ενισχύει η μία την άλλη. Αυτή όμως δεν είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέτρια ανάπτυξη όσον αφορά την παραγωγικότητα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παίζουν ε, σημαντικό ρόλο στην ε, ατυχή αυτή εξέλιξη. Έχουμε όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι ε, τα αρνητικά επιτόκια δημιουργούν περιβάλλον όπου επιβιώνουν ε, οι λεγόμενες επιχειρήσεις ζόμπι, οι οποίες δεν θα επιβίωναν αν ήταν πιο ψηλά τα επιτόκια ε, και σε κάπως πιο φυσιολογικά επίπεδα. Τέταρτον, έχουμε το σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τραπεζικού συστήματος, Πολιτικά όμως ε, δεν ε, θα γίνει αποδεκτό σε διάφορες χώρες, εκτός ε, αν γίνει περισσότερη δουλειά σε άλλες χώρες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να υπάρχουν στις χώρες αυτές. Και τέλος, η έκθεση αγνοεί τα, τις όλο και πιο σημαντικές παρενέργειες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, Μία εξαιρετικός κατάλογος των παρενεργειών αυτών είναι ε, διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ε, στρέβλωση της αξιολόγησης κινδύνου, όλο και πιο υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης, συγκέντρωση, συσσόρευση χρέους και διάφορες φούσκες. Ε, επίσης, ε, στη χώρα μου βλέπουμε ε, επίδραση στην αγοραστική δύναμη. 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς καταθέσεων ουσιαστικά είναι απώλεια τεράστια για την τελευταία δεκαετία. Επίσης, έχουμε το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και έχουμε Επίσης, ε, το άλλο αποτέλεσμα που δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε το ότι αποστέλλονται λάθος μηνύματα στον πολιτικό κόσμο, διότι οι επενδυτικές τράπεζες λένε συνέχεια ότι μπορούν και θα κάνουν περισσότερα. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι ο πολιτικός κόσμος θα κάνει λιγότερα στην περίπτωση αυτή. Ε, χρειάζονται λοιπόν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με τις τροπολογίες μας θέλουμε να καταλήξουμε σε πιο πλήρη και επιστή εικόνα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης από την QNGL. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη για το σχέδιο έκθεση που μας έστειλε και για την παρουσίαση που μόλις μας έκανε. <clears throat> Πιστεύω ότι είναι μια ικανοποιητική βάση για τη συζήτησή μας. Εμείς ε, έχουμε καταθέσει εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας 32 τροπολογίες ε, γιατί θέλουμε σε ορισμένα σημεία ε, να ενισχυθεί το περιεχόμενο της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή που δεν έχουμε απλώς μια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον κίνδυνο μιας νέας οικονομικής κρίσης τον οποίο επισημαίνει και η ίδια η ΣΥΜΠΗ και ο κύριος Ντράγκη και η κυρία Λαγκάρτ, η διαδοχός του, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ευάθυση της Ένωσης και της Νομισματικής Ένωσης και εδώ κάτι λείπει. Ο τρίτος πυλώνας, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Και έχω ακουραστεί χρόνια να ακούω εκπροσώπους διάφορων πολιτικών ομάδων να αρνούνται αυτό που προτείνει η Κομισιόν, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το οποίο αν δεν ολοκληρωθεί δεν θα έχουμε απλώς τραπεζική ενοποίηση. Και είναι η παράλληλη πορεία της μείωσης και της αμοιβεοποίησης των ρίσκων με την εφαρμογή του ίντις η θεωρία ότι πρέπει πρώτα να μηδενιστούν τα ρίσκα για να αρχίσουμε να συζητάμε την εφαρμογή του ίντις οδηγεί σε έναν μεγάλο κίνδυνο. Το δεύτερο θέμα που ε, θέλουμε να ενισχυθεί στην έκθεση είναι μια ενεργή, πιο ενεργή συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα η ε, κυρία Λαγκάρτ έχει δεσμευτεί ότι θα κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ώρα τα λόγια να γίνουν πράξη με ένα σχέδιο. Περιμένουμε άλλωστε και από την Κομισιόν την πρόταση για τον Green New Deal. Το τρίτο θέμα είναι οι συνέπειες του Brexit που απαιτούν μια πιο ενεργή παρέμβαση. Και το τελευταίο θέμα, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, είναι ότι αυτά τα χρόνια έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ οι ανισότητες, κοινωνικές και περιφερειακές, και αυτό απαιτεί να δούμε και στο νομισματικό σκέλος αλλά και στο δημοσιονομικό του σκέλος το θέμα της ευελιξίας στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά και την ανάγκη να δούμε και στο μέλλον ένα νέο σύμφωνο απασχόλησης και ανάπτυξης. Με επικοδομητικό πνεύμα αναμένουμε από τον εισηγητή τις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα μας παρουσιάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί ή να αναιρεθεί το περιεχόμενο της έκθεσης Μαυρίδη, όπως ε, θα επιχειρηθεί από ό,τι κατάλαβα από ορισμένε πολιτικές ομάδες. Thank Ευχαριστούμε. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Μαυρίδη. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ακούσαμε διάφορες απόψεις, διάφορες κατευθύνσεις που εμπλουτίζουν το διάλογο και την έκθεση αυτή. Επαναλαμβάνω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρω ισορροπημένες συμβαστικέ προτάσεις που θα επιτρέψει σε όλους μας να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 22 ή 23 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια τον Φεβρουαρίο. Διακοπή της συνεδρίασης θα ψηφίσουμε στις 5. Good afternoon. I think we are all here. Νομίζω ότι είμαστε όλοι παρόντες. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πρωτού προχωρήσουμε, να κάνουμε πρώτα μία δοκιμή. Σας παρακαλώ λοιπόν ξεκινήσουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Δοκιμή, αλλά είναι χρήσιμο και για μας να δούμε ποιοι είναι παρόντες. Λήξη της ψηφοφορίας. Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα Ε, σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, έγκριση του διορισμού του κυρίου Φάβιο Πανέτα. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. I uh, it uh, one Από ό,τι φαίνεται έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Ωραία, τώρα είναι όλα καλά. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. 51 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Διορισμός μέλους, ε, διορισμός ε, της κυρίας Ιζαμπέλ Σνάμπελ ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάλι μυστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 41 υπέρ 13 κατά, 4 αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι ορισμός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Επιτροπή και συγκεκριμένα την έγκριση του κυρίου Βέρνερ Λάνιε. Πάλι μυστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Και πάλι έχουμε... Όχι, εντάξει, όλα είναι εντάξει. Λήξη της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 10 κατά ε, τέσσερις αποχές εγκρίνεται. Okay, we move to the next uh, point. We... Προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι απαιτήσει για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Έκθεση της Λίδια Περέιρα. Ξεκινάμε με την τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 31. So sorry, I dropped the coffee. έχασα, έχισα τον καφέ μου. I am okay. No worries. That's okay. The list is safe. Okay. Εντάξει, πάντως δεν έπαθε τίποτα ο κατάλογος ε, της ψηφοφορίας. Και έχουμε φτάσει στην τροπολογία 31. ζητώ συγγνώμη για το μικρό αυτό ατύχημα. 31 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 38 είναι παρομοιότυποι. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 42. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 6, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 2 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφοφορία πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 51 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Now we are voting on the... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ψηφίσουμε τώρα για τα μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ. Άλλη μια έκθεση νομοθετική της κυρίας Περέιρα και ξεκινούμε με την ψηφοφορία για την συμβιβαστική Α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Επομένω, προχωράμε στην τελική ψηφοφορία για την πρόσθεση τη Επιτροπή όπω τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. κλίση. Ψηφίστε, παρακαλώ. Close the vote. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 50 ψήφου υπέρ, 5 2 κατά και 5 αποχές. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία για το ψήφισμα για την δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία, BEPS 2. Ξεκινούμε με την τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23 ψήφοι υπέρ, 32 κατά. Ωραία, άρα τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ακριβό ποσός και πριν απορρίπτεται. Συμβιβαστική A υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική B, Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στην συμβιβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τη συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική DA υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ζητείτε. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Για την 75. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε θα προτιμούσα. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι. E, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. δείχνουμε με την συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93, τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 105. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με 23 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 4 αποχές. Συμβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική N υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβεβαστική O. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 135 υπέρ κατά αποχές. φάνηκε ότι απερίφθη, λέει η πρόεδρος. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά όμως. Ψηφίστε για την 135. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πράγματι με 33 ψήφους κατά, 23 υπέρ και μια αποχή. Τροπολογία 141 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική T. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική U. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 160 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 164, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ζητάτε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 168. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στην 173. 173 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 173, έναρξη ψηφοφορίας. Close the vote. Πέρας. Adopted. Yes. Okay. Yeah, I they... Εγκρίνεται. Compromise XX. Συμβιβαστική XX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική X μία φορά ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Close the Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AB. ΑΒ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. κατά, ε, αποχές ε, απερίφθη, 33 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, Πέρε της ψηφορίας, απορρίπτεται, 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συμβαστική AC υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε, ψηφίστε για τη 40 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 6 αποχές. Yes. Thank you very much. So, now we vote. Και τώρα να ψηφίσουμε για τη σύσταση για την ε, ένσταση για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 39 και το 7, 7 και 9. Υπέρ. Τα ψηφίζουμε on block. 1 ε, και 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά αιτιολογικές αναφορές 1 ως 7. On block. 1, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά αρχικό κείμενο αιτιολογικής σκέψης α ως ε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε για το κείμενο διανομαστικής κλίσης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 40 υπέρ, 3 κατά, 11 αποχές. Κυρίσω τη λέξη αυτή τη συνεδρίαση και η επόμενη θα λάβει χώρα την 5η στι 7 Δεκάτου 2019 από τι 9 ω 12.30.